Eh, Συνεχίζεται η συνεδρίασή μας με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη σχετικά με το μαζικό εκτοπισμό των παιδιών στην Ιγύρια λόγω των επιθέσεων της Μπόκο Χαράμ. Ο κύριος Τέμες Μάκερ για ένα λεπτό εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα 1,2 εκατομμύρια